Ladies and gentlemen, dear colleagues. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να καθίσετε. Είναι 5 και 5 η ώρα. Καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης και τα μέλη της Υποεπιτροπής ε, Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Η πρόεδρος Μαρία Ρένα είναι μαζί μας και ο πρόεδρος είναι εδώ δίπλα μου της Επιτροπής Ανάπτυξης, ο κ. Στόβε. Δύο ανακοινώσεις ως πρόεδρος της ΑΦΕΤ. Πρώτον, θα πρέπει να υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη της ε, συνεδρίασής μας ε, και για αύριο. Δεν έχει σχόλια από πλευρά σας, πιστεύω. Δύο ανακοινώσεις που ήθελα να κάνω. Η πρώτη, να σας ενημερώσω ότι οι ψηφοφορίες για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων τριλόγων ε, δηλαδή για το μηχανισμό γειτονία ανάπτυξης και διεθνού ε, συνεργασία και για το μηχανισμό προενταξιακή βοήθειας που έχουν, έχουν προγραμματιστεί για τις 8 Οκτωβρίου και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα ε, πριν την ψηφοφορία για το βραβείο Ζαχάροφ στις, 10... στις 3 ώρα. Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία και της ΑΦΕΤ και της ΔΕΒΕ μαζί για το NDICI, ούτω ώστε να ληφθεί απόφαση έναρξη ε, τριλόγων. Οπότε είναι σημαντικό να είστε παρόντε στην ψηφοφορία στο βαθμό του δυνατού. Και η δεύτερη ανακοίνωση, πολύ σημαντική, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου με ενημέρωσε ότι δυνάμει του άρθρο 2 παράγραφου 2 παραρτήματος 7 του ιστορικού κανονισμού η διαδικασία ορισμού του Ούγκρου υποψήφιου υπετρόπου το Τζανί αναστέλλεται. Αναστέλλεται δηλαδή και η ακρόαση αύριο δεν θα λάβει χώρα. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία για την επόμενη ακρόαση. Ωστόσο, εγώ επεσήμανα στον πρόεδρο ότι το προτιμότερο είναι η ακρόαση να γίνει στις 14 Οκτωβρίου, Δευτέρα, διότι είναι η μέρα της ΑΦΕΤ ούτως ή άλλως. Αυτά ήθελα να ανακοινώσω στους συναδέλφους, συναδέλφους της ΑΦΕΤ, διότι οι συνάδελφοι της ΑΦΕΤ ε, μου στέλνουν μηνύματα από το πρωί και ζητούν εξηγήσει. Αυτά όσον αφορά τα διαδικαστικά, ναι. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε Ζερόμ Ριβιέρ, μέλος ε, της Επιτροπής αυτής. Όσον αφορά την ακρόαση, η οποία ανεστάλλει, αναβάλλεται, που δεν θα λάβει χώρα, δεν για τον εσωτερικό μας κανονισμό. Η Επιτροπή μας μήπως βρίσκεται σήμερα σε μια παράδοξη κατάσταση όπου δεν μπορεί να δώσει πολιτική γνωμοδότηση, ενώ η ε, Γιούρι έδωσε μια γνωμοδότηση πολιτική ενώ δεν έπρεπε. Ε, αντικατέστησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής που έπρεπε να δώσει. Η μόνη ε, η απόφαση που έπρεπε να λάβει η Γιούρι είναι αν, αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή όχι. Δηλαδή, και βάσει των πληροφοριών που λάβαμε φαίνεται να μπήκε στη θέση της κανονικής επιτροπής όπου θα γινόταν η ακρόαση του υποψηφίου ή των υποψηφίων επιτροπών. Θέλω την απόψή σας γι' αυτό. Καταλαβαίνω αυτό που είπατε, το σημειώνω, δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Η Επιτροπή Γιούρη αποφάσισε με πλειοψηφία και ο πρόεδρος της με ενημέρωσε ότι η υποψηφιότητα αυτή βρίσκεται σε αναστολή. Αυτά αυτή τη στιγμή. Κάποια άλλη στιγμή μπορεί να μπορέσουμε να συζητήσουμε το τι συνέβη στη Γιούρη. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε. Λυπάμαι. Εδώ τελειώνει οι ανακοινώσει του Προέδρου. Περνάμε στην κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξη και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σας καλωσορίζω όλους και όλες σε αυτή την κοινή συνεδρίαση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνουν οι παρουσιάσεις των υποψηφιωτήτων του βραβείου Ζαχάροφ για αυτή τη χρονιά από τα καινούργια ε, νεοκλεγμένα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Με το βραβείο αυτό τιμούμε ε, εξαίρετα εξαιρετικά άτομα τα οποία με κίνδυνο της ζωής τους ε, προσπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι υποψήφοι έχουν ε, αφήσει το ίχνος τους και η δουλειά τους έχει εμπνεύσει πολλούς άλλους. Αυτή είναι η αρχή της διαδικασίας για την επιλογή ε, αυτού που θα λάβει το βραβείο το 2019. Θα ακούσουμε για τους υποψήφιους σήμερα αυτούς υποψήφιους που εσείς έχετε προτείνει οι επιτροπές μας μετά θα ψηφίσουν αυτό το κατάλογο στην επόμενη συνεδρία, στην 3η 8 Οκτωβρίου ε, και τρία ονόματα θα σταλούν στην διάσκεψη των Προέδρων η οποία και θα αποφασίσει για το ποιος θα βραβευθεί απόφαση που θα ανακοινωθεί στις 24 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Το βραβείο Ζαχάροφ είναι ίσως η πιο ορατή πτυχή της, ε, του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι η μόνη πτυχή όμω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεισφέρει στι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακολουθεί το έργο των άλλων θεσμικών οργάνων ε, και προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα με δικέ του δράσει. Μέσω των, ε, των δημοσιονομικών μας αρμοδιοτήτων ε, συναποφασίζουμε για την χρήση των ποσών τα οποία προορίζονται για την προασπίση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σκοπό σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές μας τις αρμοδιότητες και τα επόμενα χρόνια. Ε, σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες συνεργασίας με τη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, σίγουρα θα λάβουμε υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και υιοθετούμε επίσης και ψηφίσματα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλές χώρες, ψηφίσματα τα οποία πραγματικά κάνουν τη διαφορά πολλές φορές. Να σας υπενθυμίσω ότι το κοινοβούλιο αυτό ε, έχει στηρίξει ανθρώπους όπως ο Ντένις Μουκβέγγε, η Νάντια Μουράτ, ε, Ράιφ Μπαντάουι και, ο τον Όλεκ Σέντσοφ. Τους στηρίξαμε για πολλά χρόνια, του στηρίζουμε για πολλά χρόνια και κυρίως όταν το χρειάζονται. Ε, νωρίτερα αυτό το μήνα με χαρά ακούσαμε, μάθαμε ότι απελευθερώθηκε ο κύριος Σέντσοφ. Θα δώσω το λόγο στον Τόμας ε, Τομπέ, τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης, ε, για να μας εισάγει στους υποψήφιους. Ευχαριστώ. Τόμας. Ευχαριστώ κύριε Μακάλιστερ. Συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά που έχω την τιμή να συμπροεδρεύω την συνεδρίαση για το βραβείο Ζαχάροφ και πρέπει να είμαστε πραγματικά όλοι περήφανοι που έχουμε την ευκαιρία να είμαστε εδώ. Το βραβείο Ζαχάροφ δεν είναι μια διαδικασία τυπική. Είναι μια ευκαιρία να φωτίσουμε το, τη δουλειά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές ανθρωπινών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Και αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο εντός του οποίου εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζουμε τις εξαιρετικές, την εξαιρετική προσφορά ε, ανθρώπων στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας και τους δίνουμε θάρρος και κουράγιο για την ε, προσήλωσή τους. Ε, η παρουσίαση των πέντε υποψηφίων θα γίνει αλφαβητικά. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους υποψηφίους μπορείτε να δείτε και το φυλάδιο το οποίο έχει ε, επισυναυθεί στο φάκελο που έχετε λάβει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την παρουσίαση των υποψηφίων. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε προβλέψει 10 λεπτά το πολύ για κάθε υποψηφιότητα. Και γι' αυτό εμπιστευόμαστε, σας εμπιστευόμαστε ότι θα τηρήσετε αυτόν τον ε, κανόνα γιατί θέλουμε να κάνουμε και μια ανταλλαγή απόψεων στη συνέχεια διάρκειας 15 λεπτών. Να, σας δώσω τώρα το λόγο. Ξεκινάμε με την πρώτη υποψηφιότητα. Είναι η Μαριέλ Φράνκο, ο αρχηγός Ραόνι και η Κλοντλής Σίλβαντο Σάντος, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Υποψηφιότητα που υπευλήθη από τους σοσιαλιστές και την ΚΟΕ. Θα ξεκινήσουμε με, την, ε, με ένα σύντομο βίντεο και στη συνέχεια θα ακούσουμε τις παρεμβάσεις ε, της κυρίας Ιζαμπέλ Σάντος και της κυρίας Μαρίσα Ματίας από τους σοσιαλιστές και την ΚΟΕ αντίστοιχα. Ξεκινάμε με το βιντεάκι και ε, ελπίζουμε να λειτουργήσει και τεχνικά.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 Να ακούσουμε την κυρία Ισαμπέλ Σάντο από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Είναι μεγάλη τιμή μας ε, εκ μέρους της ομάδας των σοσιαλιστών να υποβάλουμε την κοινή αυτή υποψηφιότητα Μαριελ Φράνκο, Φιλάρχου Ραονί και Κλαουντελίσε Σίλβα Ντουσάντος και είναι τιμή που μπορούμε αυτή την παρουσία να την κάνουμε στα πορτογαλικά, είναι η γλώσσα η οποία τους ενώνει. Αυτή η κοινή υποψηφιότητα αντιπροσωπεύει της, ε, τη φωνή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος στην Βραζιλία και κυρίως στην Αμαζονία. Ο Ραόνι είναι γνωστός ως φύλαρχος. Ραόνι είναι... Ε, οικολόγος στην Βραζιλία, είναι χαρισματικός ηγέτης ε, του λαού της φυλής των Καγιάπο ε, που ζει στο, στην περιοχή του Ματογκρόσο στην Αμαζονία και κατά το μήκος του ποταμού Τσίνκου. Εδώ και 40 χρόνια κάνει μια εκστρατεία, μια σταυροφορία θα λέγαμε να σώσει το περιβάλλον στην Αμαζονία. Ε, έχει ξεκινήσει ένα αγώνα για την προστασία της, ε, των τροπικών δασών και έχει διακινδυνεύσει τη ζωή τους αυτό. Η Κλαουντελίση Σίλβα του ε, είναι μια ε, οικολόγος στην Βραζιλία, ακτιβίστρια, έγινε ακτιβίστρια μετά τη δολοφονία της κουνιάδας και του αδελφού του που πολεμούσε εναντίον των παράνομων ξυλοκόπων πάνω από 1.500 άτομα μεταξύ του 2000 και του 2017 δολοφονήθηκαν σε 50 χώρες του κόσμου επειδή ακριβώς προσπάθησαν να προασπίσουν ε, την ε, χλωρίδα, το νερό και τη γη τους. Είναι αδιανόητο άνθρωποι να δολοφονούνται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την προστασία ενός ε, κοινού αγαθού. Η Μαριέλ Φράνκο ε, μετά το θάνατό της, μετά θάνατον. Ε, γεννήθηκε το 1979. Ε, έχασε τη ζωή της τον ε, φέτος, το Μάιο. Ήταν φεμινίστρια, ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανοιχτά. Ε, επίσης ήταν θύμα της ε, ε, αστυνομικής βίας. Ε, ήταν δημοτική σύμβουλος στο Δήμο του Ρίο Ντετζανέιρο. Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια φαβέλα του Ρίο και εργαζόταν από παλιά στην προστασία των, ανθρωπι... των δικαιωμάτων των γυναικών, των νέων και των ΛΟΑΔ. Στις 14 Μαΐου 2018, γυρνώντας με το αυτοκίνητο από μια ομιλία της, ε, δολοφονήθηκε μαζί με τον οδηγό της ε, από δύο άτομα τα οποία διέφυγαν με ένα όχημα τον Μάρτιο του 2019 δύο πρώην αστυνομικοί συνελήφθησαν και κατηγορούνται με τη δολοφονία της. Σύμφωνα με την ομάδα Gay της Μπαϊά, 420 άτομα της κοινότητας ΛΟΑΤ στη Βραζιλία έχουν χάσει τη ζωή τους από ανθρωποκτονίες ή ε, αυτοκτόνησαν το 2018 κατόπιν ε, πράξεων ομοφοβικών. Ε, οι απειλές ε, αυξάνονται και εντείνονται εναντίον της ζωής και της ακαιρεότητας των ακτιβιστών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΛΟΑΤ, αλλά και δημοσιογράφων. Η Βραζιλία είναι η χώρα, η πιο επικίνδυνη χώρα για τη ζωή ακτιβιστών, τέτοιων ακτιβιστών, αλλά και ακτιβιστών φυλών ε, που προασπίζουν το περιβάλλον. Η Αμαζονία, μάλιστα, είναι η περιοχή της Βραζιλίας που πιο πολλές δολοφονίες έχουν εμφανιστεί, έχουν καταγραφεί το 80% του συνόλου των θανάτων, σύμφωνα με την Witness. Και μάλιστα μπορεί οι δολοφονίες να είναι ακόμα περισσότερες. Το 2018 160 ακτιβιστές του περιβαλλοντικοί οικολόγοι ακτιβιστές έχαναν τη ζωή του ε, η, ο κλάδος ε, της, ε, των, της εξόριξης και το, και η βιομηχανία ε, αποψήλωση των δασών είναι η κύρι, τα κύρια αίτια οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται ε, στο πεδίο δράσης τέτοιων ανεύθυνων επιχειρήσεων, εταιριών, ε, οι οποίες χρησιμοποιούν πληρωμένους δολοφόνους. Και επειδή δεν αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα, δημιουργείται ατιμορρησία. Ο, το περιβάλλον έχει γίνει ε, το νέος το νέο πεδίο μάχη ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το να απονείμουμε το βραβείο Ζαχάροφ σε αυτά τα άτομα είναι ένα τρόπο να προασπίσουμε το περιβάλλον αλλά και του υπερασπιστέ του, του περιβάλλοντος, φέρνοντάς τους στο κέντρο τη πολιτική μα ατζέντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Μαρίζα Ματίας από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η Βραζιλία συνταράσσεται και αυτή η υποψηφιότητα είναι σημαντική. Σε αυτή την κοινή πρόταση προσπαθούμε να δώσουμε φωνή σε τρία άτομα τα οποία έχουν συνεισφέρει με τρόπο εξαιρετικό στην, ε, στην των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η κατάσταση στη Βραζιλία είναι πολύ ανησυχητική, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτήν, ιδιαίτερα στην Αμαζονία. Εκεί θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση ε, στα προβλήματα που έρχονται από την κλιματική αλλαγή. Με τον ε, Μπολσονάρο ε, η κρατική η πολιτική οδηγεί στην καταστροφή του πλανήτη. Θα πρέπει να προστατεύσουμε την Αμαζονία από τις μεγάλες βιομηχανίες που την εκμεταλλεύονται αλλά και να προστατεύσουμε τους ντόπιου πληθυσμούς και τις φυλές που ζουν εκεί η πολιτική βία η οποία οδηγεί, οδήγησε στην ε, πράξη, ε, στην φυλάκιση του Λουάντα Σίλβα και στην απομάκρυνση της προηγούμενης ε, προέδρου πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το χωρίς όρους διεθνές εμπόριο δημιουργεί ε, πολλά προβλήματα ε, και στις, ε, στους ντόπιους πληθυσμούς αλλά και στους Ευρωπαίους παραγωγούς. Επίσης δημιουργεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα. Τρία άτομα λοιπόν οι υποψήφοι μας που έχουν ξεχωρίσει ο καθένας για την προάσπιση διαφορετικών αξιών. Προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προάσπιση του περιβάλλοντος. Όλα αυτά έχουν σχέση με τις εγγύσεις που πρέπει να δώσουμε στι μελλοντικέ στις Αυτοί είναι λοιπόν οι τρεις μας Υποψήφιοι Η Μαρία Φράνκο ε, προσπάθησε να προασπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, των μαύρων, ε, των ΛΟΑΤ και των φτωχών. Ήταν η ίδια μαύρη, ε, αμφιφιλική ε, και δημοτική σύμβουλος. Από πιο παλιά είχε ξεκινήσει τον αγώνα της, ε, αλλά για αρκετά χρόνια ήταν δημοτική σύμβολο στο Ρίο Τζανέιρο ε, και είχε καταγγείλει επανειλημμένω ε, παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δύο εβδομάδε πριν δολοφονηθεί η Μαριέλ είχε οριστεί συντονίστρια και ησυχήτρια για την αστυνομική βία στο Ρίο Τζανέιρο μια έκθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ε, ε, οι διαδικασίες μετά τη δολοφονία της ε, δεν ήταν ορθές, έχουν καταγγελθεί και βρίσκονται υπό έλεγχο. Η Κλαουντελή Σίλβα Σάντους έχει αγωνιστεί εναντίον της, ε, της παράνομης ξύλευσης ε, και των παραγωγών ε, κάρβουνου που καίνε τα δάση στη Βραζιλία. Ο αδελφός της και η σύζυγός αυτού είχαν δολοφονηθεί λόγω του ότι ήταν ακτιβιστές στην, στα τροπικά δάση της Αμαζονίας. Έξι μήνες μετά η η ίδια ε, ξεκίνησε να προσπάθησε να μετατρέψει τον, τον τοπικό αγώνα σε εθνικό αγώνα στην ε, Βραζιλία και ε, συγκάλεσε μια ένα διεθνέ συνέδριο στη Βραζιλία μάλλον ναι, στη Βραζιλία για την ε, προσ... προάσπιση της γης και των δασών της Αμαζονίας. Από την άλλη μεριά, ο φύλαρχος Ραόνι είναι εμβληματική φιγούρα. Είναι ένας από τους μεγάλους ηγέτες ε, της Αμαζονίας. Είναι σχεδόν 90 ετών και έχει συμπληρώσει πολλές δεκαετίες αγώνα υπέρ των δικαιωμάτων ε, των ε, τοπικών φυλών και υπέρ του περιβάλλοντος. Ε, βοήθησε στην συνειδητοποίηση της ανάγκης να προστατευθούν. Η δράση του οδήγησε στη δημιουργία μιας, ε, ε ενός μιας προστατευμένης έκτασης 180.000 τραγωνικών χιλιόμετρων στην Αμαζονία. Ε, αυτή τη στιγμή ο Μπολσον, ε, πολλές ε, φυλές ε, της Αμαζονίας φοβούνται ότι ο Μπολσονάρο με την πολιτική του θα οδηγει στην καταστροφή τους. Αυτές λοιπόν οι τρεις μορφές ε, αποτελούν και αντιπροσωπεύουν την ουσία του βραβείου Ζαχάροφ. Δίνουν φωνή σε ανθρώπους που δεν θα είχαν φωνή αλλιώς. Η Μαρία Ελφράνκο δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας προφανώς. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και το δικό της έργο. Είμαστε περήφανοι που του έχουμε προτείνει ω υποψήφιου. Ευχαριστώ. So, thank you. Ωραία. Και με αυτό ολοκληρώσαμε την παρουσίαση του πρώτου υποψηφίου, της πρώτης υποψηφιότητας. Μιλάμε πλέον για το δεύτερο υποψήφιο που είναι ο Αλεξέη Ναβαλνή που έχει υποβληθεί ως υποψηφιότητα από το ΕΛΚ. Θα δούμε ένα βίντεο. Мы вместе, и мы победим!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 and continue to erupt. Pressure grows on Putin to change his evil ways and end his autocratic rule. Thank you. Now I give the... Ευχαριστώ. Να ακούσουμε την ε, κυρία Σάντρα Καλινέτε. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Το Ευρωπαϊκό Λογικό Κόμμα υποβάλλει την υποψήφια του Αλεξέη Ναβάλνη, ενός πολιτικού ηγέτη της Ρωσίας, για την απονομή σε αυτόν του βραβείου Ζαχάροφ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο κ. Ναβάλι μπορεί να συμβάλλει στον αγώνα που γίνεται στη Ρωσία για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η μεγάλη υποστήριξη και η μεγάλη πορεία του Ναβάλι, παρά την καταστολή που έχει δεχτεί από τις αρχές, ο ίδιος, οι υποστηρικτές του, οι συγγενείς του, δείχνει την προσήλωσή του σε αυτές τις αξίες. Ο Λαμβάλνη αναγνωρίζεται διεθνώς αλλά και ε, μέσα στη χώρα του ως ε, πραγματικός ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Ρωσία. Από το 2008 ο Λαμβάλνη είναι αγωνιστής ενεργός κατά της διαφθοράς στον ε, κρατικό μηχανισμό και στις, κρατικά, ε, στις επιχειρήσεις κρατικής ιδιοκτησίας. Ο οργανισμός του που, ε, θεσπίστη, που δημιουργήθηκε το 2011 αποκαλύπτει περιπτώσεις διαφθοράς και νεποτισμού. Το κανάλι του στο YouTube είναι ένα από τα κανάλια με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στη Ρωσία, με πάνω από 3, 3 ε, εκατομμύρια ακολούθους. Το 2013 ο Ναβάλνη ήταν υποψήφιος ε, για δήμαρχος της Μόσχας και κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Έκτοτε αντιμετωπίζει συνεχείς πιέσεις από τις αρχές και του έχει απογορευτεί η συμμετοχή του σε εκλογές τοπικές, περιφερειακές και προεδρικές. Έχει ε, ε, πάνω από 300 ε, μέρες ε, περάσει σε φυλακές ε, έπειτα από παραβίαση του εκλογικού νόμου και του νόμου περί διαμαρτυριών. Από το 2016 πάνω από 3.000 άνθρωποι ε, έχουν κρατηθεί. Ωστόσο, ε, λόγω της ε, στρατηγικής του Ναβάλνη για την έξυπνη τακτική να υποστηριχθούν υποψήφοι αντιπουτινικοί στέφθηκε με επιτυχία. Ε, έτσι εξελέγησαν πάρα πολύ τοπικοί ε, δημοτικοί σύμβουλοι, 13 συγκεκριμένα. Σας καλούμε λοιπόν να υποστηρίξετε αυτή την ε, υποψηφιότητα του Αλεξέη Ναβάλνη για το βραβείο Ζαχάρεφ και με αυτόν τον τρόπο να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην κοινωνία των πολιτών της Ρωσίας ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφού γκραζόμαστε τις φωνές ε, της νέας γενιάς ε, της Ρωσίας που θέλουν αλλαγή και μια ε, εναλλακτική στο υπάρχον καθεστώς της Ρωσίας. Ευχαριστώ. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Γκάλερ. Συναδελφοί, Πράγματι η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερο γείτονά μας στην Ανατολική Ευρώπη και ένα διαρκέ πρόβλημα. Πιστεύω ότι για να υπέρθει αλλαγή στη Ρωσία και για να υποστηρίξουμε όσους θέλουν να φτιάξουν μια δημοκρατική κοινωνία σε αυτή την χώρα είναι να υποστηρίξουμε τον αγώνα τους και την κοινωνία των πολιτών στη χώρα αυτή είτε το γνωρίζετε είτε όχι, όταν δημιουργήθηκε το βραβείο Ζαχάροφ το 1988, το όνομα δόθηκε λόγω ενός Ρώσου βραβευθέντος, αλλά ουδέποτε βραβεύθηκε άλλος Ρώσος στη συνέχεια. Και δυστυχώς ε, πρέπει να είναι κάποιος από μια χώρα που η δημοκρατία και η ελευθερία του λόγου είναι περιορισμένη όπως και στη Ρωσία, αλλά πρέπει να πούμε ότι η κατάσταση αυτή επιδρά ε, στη ρωσική κοινωνία λόγω της κακής κυβέρνησης εκεί και έχουμε να κάνουμε με την επιθετικότητα και στις εξωτερικές σχέσεις επίσης. Για να βρεθεί ένας τρόπος λοιπόν να ενθαρρύνουμε τη ρωσική κοινωνία να εκφράσει τις επιθυμίες της για αξιοπρεπή ζωή και πιο πλουραλιστική κοινωνία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς ε, που είναι γνωστοί, που βροντοφωνάζουν τα όσα λαμβάνουν χώρα σε αυτή τη χώρα και εμείς ε, προσδορίσαμε, εντοπίσαμε τον Αλεξέη Ναβάλνη ως ε, μια σημαντική προσωπικότητα που μέσω ομιλιών και δραστηριοτήτων απέδειξε ότι μπορεί να διατυπώσει την επιθυμία ενός ολένα αυξανόμενου μεριδίου της κοινωνίας ε, στη Ρωσία. Πιστεύω ότι αυτός είναι και ο μόνος τρόπος ε, ώστε να φέρουμε πιο κοντά μας στη Ρωσία και πιο κοντά στους άμεσους γείτονές της ε, που ακόμη φοβούνται τη χώρα αυτή. Πιστεύω οι Ρώσοι δεν αξίζουν τέτοια αντιμετώπιση, δεν τους αξίζει να τους φοβούνται οι άλλοι για να βρουν λοιπόν το δρόμο προς περισσότερη δημοκρατία και πλουραλισμό στη Ρωσία, πρέπει να υποστηρίξουμε ανθρώπους όπως τον Αλεξέη Ναβάλνη. Εμείς λοιπόν ως ΕΛΚΑ τον υποστηρίζουμε για να λάβει το γραφείο Ζαχάροφ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ που δεν ξεπεράσετε το χρόνο ο, για το δεύτερο υποψήφιο. Ο τρίτος υποψήφιος είναι μια ομάδα ε, μαθητών από την Κένια που ονομάζεται The Restorers. Ε, τους, ε,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 Ευχαριστούμε. Δίνουμε το λόγο στην κυρία Σίτα Κανκού. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό που ήθελα να πω για τους restorers, θέλω να σας παρακαλέσω να σταθείτε δίπλα μου. Να συνδράμουμε τα κορίτσια που φωνάζουν βοήθεια. Πιστεύω ότι με αυτή την πρωτοβουλία που έχω αναλάβει ομάδα ανθρώπων στην ΚΕΝΕ και μπορεί να επεκταθεί παγκοσμίω να επεμβαίνουμε πριν αρχίζουν να κλαίνε τα κορίτσια. Εγώ όταν με ακροτηρίασαν δεν ήρθε κανένας και αυτό με πλήγωσε περισσότερο. Έχουμε λοιπόν τώρα αυτή την επιλογή. Μιλάμε για 7 κορίτσια το λεπτό. 500.000 θύματα που ζουν στην Ευρώπη. Τις ονομάζω επιβιώσασες, διότι κάθε μέρα πρέπει να ανακτήσεις την αυτοπεποίθησή σου και εγώ ακόμα αγωνίζομαι και καθημερινά, ξέρεις ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλους ανθρώπους. Πώς μπορείς λοιπόν να τους βοηθήσεις είναι αυτό που σε απασχολεί. Όταν σε ακροτηριάσουν όταν είσαι παιδί, δεν χάνεις απλά ένα ευαίσθητο προσωπικό κομμάτι του σώματός σου, αλλά και κάτι άλλο το οποίο δεν μπορείς να ανακτήσεις ποτέ. Το πώς θα ήταν το σώμα σου και πώς θα ήταν η ζωή σου αν δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο χάνεις ε, τη γέφυρα που σε συνδέει με τους γονείς σου, πώς θα μπορέσεις να εμπιστευτείς οποιονδήποτε ξανά. Δεν τους εμπιστεύεσαι τους γονείς σου ξανά. Κάτι απαραίτητο για ένα παιδί. Δεν υπάρχει κανένα στον οποίο να μιλήσεις, στον οποίο μπορείς να μιλήσεις. Είναι ταμπού, απαγορεύεται να συζητήσεις γι' αυτό. Αυτό που μου αρέσει λοιπόν σε αυτή την πρωτοβουλία, σε αυτή την εφαρμογή, είναι ότι αυτό που νιώθεις ε, ε, μπορεί ελεύθερα να σε βοηθήσει να δράσεις χωρίς να σκέφτεσαι. Δεν φοβούνται τα κορίτσια ε, όπως φοβούνται να μιλήσουν στη μάνα τους. Εμένα ε, μου πήρε 20 χρόνια για να πω σε οποιονδήποτε, να το πω σε οποιονδήποτε. Οπότε παρακαλώ υποστηρίξτε αυτά τα κορίτσια. Η υποστήριξη δεν είναι μόνο για αυτές. Είναι για να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Τα κορίτσια αυτά κάθισαν, αποφάσισαν να καθίσουν και να κλάψουν θα μπορούσαν να ε, είχαν καθίσει κάτω και να κλάψουν και να μην κάνουν τίποτα, αλλά αποφάσισαν να λάβουν δράση. Και κάποιοι άνθρωποι κάνουν κάτι τέτοιο στην Αφρική. Αυτό μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και εδώ. Όχι μόνο για αυτού του είδου τη βία που είναι πολύ συγκεκριμένη, αλλά και για άλλου τύπου βία. Και όταν θα απονεμηθεί το βραβείο Ζαχάροφ, τι γίνεται στη συνέχεια, όλοι είμαστε ικανοποιημένοι ε, και πάμε σπίτι μας μετά ή θέλουμε να συνεχίσουμε μετά να κάνουμε κάτι μέσω αυτού του κοινοβουλίου ανεξαρτήτως της πολιτικής ομάδας από την οποία προερχόμαστε μπορούμε να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα εγώ με τους restorers αυτό θέλω να κάνω να τους βοηθήσουμε αλλά και να συνεχίσουμε σε αυτό το κοινοβουλίο να βοηθήσουμε τα κορίτσια αυτά να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τα κορίτσια αυτά γι' αυτό λέω ότι αυτό το θέμα δεν έχει να κάνει με το ECR ούτε τις πολιτικές ομάδες, τα πολιτικά κόμματα. Όταν ένα πεντάχρονο και εγώ πέντε χρονών ήμουν, φωνάζει βοήθεια. Δεν έχει σημασία ποιο θα έρθει. Απλά πρέπει να έρθει κάποιο. Και εγώ ήθελα μόνο τη μητέρα μου. Και αυτό θέλουν και αυτά τα κορίτσια. Σα ευχαριστώ για την υποστήριξή σα. Thank you. Uh, was Ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η τρίτη υποψηφιότητα. Περνάμε στην τέταρτη υποψηφιότητα. Ilham Tohti. Έχει υποβληθεί από την ομάδα Renew Europe τον Φιλίπ Μπενιόν, τον Ilhan Κιουτσούκ, τον Reinhard Beauty και 58 άλλα μέλη. Θα ξεκινήσουμε με ένα βίντεο.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 我唯一的牵挂就是母亲和孩子们。Thank you, now I give, uh... Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κιτσουκ. Δυστυχώς η Κίνα συστηματικά παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία της έκφρασης, ε, του συνεταιρίζεστε, τα θρησκευτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Οι κινέζικες αρχές μάλιστα ε, κάνουν το ίδιο και ιδιαίτερα με την ε, εθνοτική ομάδα των Ουιγούρων. Η έχουν ανοίξει στρατόπεδα επανεκπαίδευσης όπου γίνεται πλήση εγκεφάλων και πολλές φορές και βασανιστήρια στους Ουιγούρους. Αυτό είναι τρομακτικό. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί. Η ομάδα Renew Europe μαζί με συναδέλφους άλλων πολιτικών ομάδων αποφάσισαν λοιπόν ε, να προτείνουν τον καθηγητή Ιλχάμ Τόχτη για το βραβείο Ζαχάροφ 2019. Ο κ. Στόχτη δεν είναι απλώς ο πιο σεβαστός διανοούμενος Σουηγούρος στον κόσμο. Ε, είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί ειρηνικά να συμφιλιώσει τους Σουηγούρους με τους Κινέζους. Και αυτό το λόγο όμως έχει γίνει νούμερο ένα στόχος της Κίνας. Ε, η δική του συμπεριφορά και προσέγγιση είναι ήπια. Έχει κατηγορηθεί όμως για αποσχιστικές ε, δράσεις πάνω από ένα εκατομμύριο Ουιγούρ βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα στρατόπεδα επανεκπαίδευση και η δράση του κυρίου Τόχτη είναι φωνή όλων αυτών. Το 2016 ξεκινήσαμε να τον προτείνουμε για το βραβείο Ζαχάροφ και επιμένουμε γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η φωνή θα πρέπει να ακουστεί. Ο κύριος ε, Φίλιπ Μπενιόν έχει το λόγο από το Ευχαριστώ. Ο Ήλχαμ Ταχτή για πάνω από δύο δεκαετίες προσπάθησε να ενισχύσει και να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ Κινέζων και Ουιγούρων. Προσπαθούσε για τη συμφιλίωση και όχι την απόσχηση. Ο Τόχτη ανήκει σε μια νέα γενιά ε, συγγραφέων που κινδυνεύουν, που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής για να περάσουν τα μηνύματά τους. Ωστόσο, ε, προσπαθεί, ε, δραστηριοποιείται σε μια χώρα όπου η ελευθερία έκφρασης ε, δεν υπάρχει. Μια δίκη παροδία τον οδήγησε σε ισόβια κάθριξη. Δεν έχει δει την οικογένειά του. Η οικογένειά του δεν έχει καμία πληροφορία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος αυτό. Αυτό είναι αδιανόητο σε μια δημοκρατία. Οι Ουιγούροι δέχονται πρωτοφανή καταστολή τα τελευταία χρόνια από τους Κινέζους λόγω της εθνικής τους ταυτότητας και των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων. Από το 2017 αυθαίρετα κρατούνται εκατομμύρια Ουιγούροι σε στρατόπεδα επανεκπαίδευσης όπου καλούνται να καταγγείλουν την ε, εθνική τους ταυτότητα και να δηλώσουν την ε, προσήλωσή τους και τη δέσμευσή τους στην κινέζικη κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βραβευτεί ο Ιλχαμ Τοχτή λόγω της δραστηριότητάς τους και της σχέσης του, της ε, δραστηριότητας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για μια προσπάθεια να αποκρουστεί η κρατική βία εναντίον θρησκευτικών ε, μειονοτήτων. Πρόκειται για ένα αυταρχικό κράτος που προσπαθεί να καταστήλει ένα μη βίαιο θρησκευτικό κίνημα. Για την δράση του ο καθηγητής Τόχτη έχει βραβευτεί πολλαπλώς. Έχει επίσης υπάρξει και στο παρελθόν υποψήφιος για το βραβείο Ζαχάροφ και δυστυχώς η κατάσταση από τις τελευταίες υποψηφιότητες του έχει επιδεινωθεί. Πρόκειται για ένα παράδειγμα ε, των όσων ε, πρέσβευε και ο Ζαχάροφ, ο Αντρέη Ζαχάροφ. Γι' αυτό και θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω να στηρίξετε την υποψηφιότητα αυτή. Ευχαριστώ ο κύριος Μπιούτι για τους πράσινους. Ζαχάροφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία σκέψης για εξαιρετικές προσωπικότητες που υπερασπίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ελευθερία σκέψη σε όλο τον κόσμο. Ο καθηγητή Τόχτη υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ακαδημαϊκή ελευθερία με τρόπο χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνικό μέσω των ε, γραπτών και διδασκαλιών του ενθαρρύνει τους άλλους να μοιραστούν τις ίδιες σκέψεις, να δεχθούν ο ένας τον άλλο και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο υποστηρίζει την ελευθερία ανταλλαγή ιδεών στο, στο Πανεπιστήμιο όπου εργάζεται και πέραν αυτού για την πρόθεση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η απονομή του βραβείου Ζαχάροφ στον καθηγητή Τόχτη θα σήμαινε ότι η ειρηνική ανταλλαγή ιδεών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μια ειρηνική κοινωνία και ότι ο διάλογο και ο σεβασμό είναι σημαντικά θεμέλια για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίω. Θα ήθελα επίση να προσθέσω μια απλή αλλά πικρή σκέψη και πρόταση. Οι Ουιγούροι στο Τσιαντζάν βιώνουν το χειρότερο αστυνομικό κράτος, αστυνομοκρατούμενο κράτος που γνωρίζει ο κόσμος σήμερα. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν τους υπερασπιστεί, ποιος θα τους υπερασπιστεί με τον Ινχαμ και την υποψηφιότητά του, τιμούμε την προσωπικότητα που εκπροσωπεί το αυστηρότερη και ειρηνικότερη φιλοδοξία των ανθρώπων αυτών. Thank you. That... Ευχαριστώ. Ήταν η τέταρτη υποψηφιότητα. Περνάμε στην πέμπτη και τελευταία υποψηφιότητα, Ζων Βίλης και Μαριέλ Φράνκο, που προτείνονται από την ομάδα των Πρασίνων και που θα μας τους παρουσιάσει η κυρία Νόεμαν. Ας δούμε όμως πρώτα ένα σύντομο βίντεο.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 Ευχαριστώ. Η κυρία Χάνα Νόημαν, εκ μέρους των ε, Πρασίνων. Συνάδελφοι, η Μαριέλ Φράγκο ήταν 11 χρονών όταν ως πλανόδια πολίτρια χρειαζόταν να πουλήσει πράγματα στο δρόμο. Τελείωσε όμως το σχολείο, τελείωσε το πανεπιστήμιο και συνέχισε να υπερασπίζεται τους άλλους που ζούσαν στις φαβέλες του Ρίο Τεζανέρο, όπως και εκείνη. Εξελέγει δημοτική σύμβουλος του Ρίου και αντιμετώπισε απειλές και ομοφοβία. Στις 14 Μαρτίου του 2018 δολοφονήθηκε εκείνη και ο οδηγός της. Για εμένα η Μαριόελα Φράνκο ε, αποτελεί ένα σύμβολο της πολυμορφίας της βραβλίας. Ήταν αφρολατίνα, ήταν ε, μητέρα, ήταν γυναίκα, ήταν λεσβία, ήταν γεμάτη πάθος και ήταν μόλις 39 χρονών όταν δολοφονήθηκε. Ο Ζιν Willis από την άλλη μεριά είναι ακόμα εν ζωή. Όμως είναι ο πρώτος ε, ανοιχτά γκέι βουλευτής του Βραζιλιάνικου Κοινοβουλίου και εκείνος ε, αγωνίζεται για την ΛΟΑΔ κοινότητα. Και λόγω της ε, δουλειάς του και της δραστηριότητάς του επίσης δέχτηκε απειλές για τη ζωή του, κατά τη ζωή του. Τα τελευταία χρόνια μπορούσε να φύγει από το σπίτι του μόνο με σωματοφύλακε. Στην ουσία το σπίτι του έγινε η φυλακή του. Και όλα αυτά διότι με πάθος υπερασπιζόταν τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ και άλλων μειονοτήτων στη Βραζιλία. Επειδή μιλούσε και επειδή δεν σιωπούσε. Και παρά το γεγονός ότι δεν ήθελε ποτέ να φύγει στην εξορία, αναγκάστηκε φέτος να, να φύγει. Και Όσοι γνωρίζετε ακτιβιστές στην εξορία, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να κάνει κανείς ένα τέτοιο βήμα. Μπορεί στη Βραζιλία τα γκέι ζευγάρια να έχουν ε, δικαιώματα σε γάμο και στην υιοθεσία, όμως αυτό δεν αρκεί για να τους προστατεύσει από ενέργειες βίες, που πολλές από αυτές ενθαρρύνονται ακόμη και από τον ίδιο τον ε, πρόεδρο πολλές φορές. Δυστυχώς ε, η Βραζιλία έχει ένα θλιβερό ρεκόρ είναι η χώρα στην οποία γίνονται οι περισσότερες δολοφονίες ομοφιλοφίλων. Πάνω από ένας άνθρωπος την ημέρα δολοφονείται στη Βραζιλία λόγω των, ε, της, των ερωτικών του προτιμήσεων. Ο Ζαν Βίλης λοιπόν και η Μαριέλ συμβολίζουν τον αγώνα τόσων ανθρώπων που ε, υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και που αγωνίζονται κατά της ε, βίας και των διακρίσεων. Για εκείνους που το κάνουν όχι μόνο στην Βραζιλία, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κοινότητα ΛΟΑΔ αντιμετωπίζει διώξεις και βία. 72 χώρες σήμερα συνεχίζουν να ποινικοποιούν τη σεξουαλικότητα και συνάδελφοι, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Η Μαριέλ Φράγκο και ο Ζιν Βίλη ήταν ε, πολιτικά όντα, δεν κάναν τίποτα άλλο. Ήταν πολιτικοί. Προσπάθησαν, προσπαθούσαν να καταπολεμήσουν την ε, βία, ε, υπερασπίζονταν τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια. Και παρόλα αυτά η Μαριέλ είναι νεκρή και ο Ζαν Βιλής χρειάστηκε να φύγει στην εξορία. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζονται εκστρατείε λάσπη και κατασυγκοφάντηση εναντίον του. Και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Οι πράσινοι και 43 άλλοι ευρωβουλευτέ έχουν προτείνει τον Ζαν Βίλη και τη Μαρία Φράγκο για το φετινό βραβείο Ζαχάροφ, γιατί θεωρούμε ότι οι φωνέ του αξίζει να ακουστούν. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να, να προσπίσουμε τον αγώνα του και πιστεύουμε ότι η δουλειά του πρέπει να υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ είναι αναμφισβήτητα ανθρώπινα δικαιώματα. Και γι' αυτό είναι πλέον καιρό το βραβείο Ζαχάροφ να απονεμηθεί σε ανθρώπου που εκπροσωπούν την κοινότητα ΛΟΑΔ και που υπερασπίζονται τα ίσα δικαιώματα. Όπω έκαναν. Ε, όπως έκανε η Μαριέλ Φράγκο στη διάρκεια της ζωής της και όπως κάνει ακόμη και σήμερα ο Ζαν Βίλης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ συνάλφοι για αυτές τις υποψηφιότητες. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Αρένα ε, που θα προεδρεύσει τις ανταλλαγές απόψεων. Ωραία. Ο λόγος είναι σε εσά πλέον. Κυρία Μαρκετάκη θέλει το λόγο ε, και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Ε, μέχρι τις 6.30 έχουμε χρόνο καθένας και κάθε μία από τους ε, υποψήφιους που παρουσιάστηκαν αξίζει προφανώς ε, το βραβείο Ζαχάροφ. Και μάλιστα όχι μία, αλλά δέκα, εκατό και χίλιες φορές ο καθένας. Αλλά ας δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο κόσμος. Η κατάσταση του κόσμου μας δείχνει σήμερα ότι η πιο ισχυρή δικτατορία, η πιο τεχνολογική, η πιο μοντέρνα δικτατορία και συνεπώς η πιο τρομακτική δικτατορία. Η δικτατορία που δείχνει ενδεχομένως τι θα είναι η δικτατορία του αύριο, ξέρουμε ότι είναι το κινέζικο καθεστώς. Το καθεστώς αυτό είναι τόσο ισχυρό στην διεθνή σκηνή και η κινέζικη οικονομία είναι τόσο ισχυρή που εκφοβίζει. Αυτό δεν αποτελεί δική μου ερμηνεία, είναι γεγονός. Εκφοβίζει τις περισσότερες, αν όχι όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου. Σήμερα, το ακούσαμε προηγουμένως, μπορούν να πάρουν ελεύθερα θέση για τα θέματα καταπίεσης στην Κίνα, όχι μόνο των Ιγούρων, αλλά και άλλων πολιτών. Εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας. Είμαστε το μόνο βαρύνον διεθνές όργανο που με ελευθερία μπορεί να τοποθετηθεί περί της απουσίας ελευθεριών στην Κίνα. Αν δεν το κάνουμε σήμερα, αυτή τη χρονιά, που είναι η χρονιά του Χονγκ Κονγκ και βέβαια της καταπίεσης των Ιγούρων, θα χάσουμε, ε, θα μάλλον υπολοιπόμαστε των καθηκόντων μας. Γιατί έχουμε τα μέσα να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ. Θα σε ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω το λόγο στην Τζούγκο Βίλτσε. Συγγνώμη για την κακή προφορά. Εγώ είμαι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα φυσικά να δίναμε το γραφείο Ζαχάροφ σε όλους τους υποψηφίους. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρουσίαση όλων, αλλά πρέπει να επιλέξουμε έναν. Ε, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας τη δική μου εμπειρία. Πριν από 30 χρόνια και πάνω οι Λιθουανοί ενώθηκαν στο κίνημα ανεξαρτησίας για να απαιτήσουν ελευθερία από την Σοβιετική Ένωση. Θέλαμε να ξεφορτωθούμε τον απολυτερχική δικτατορία του Κρεμλίνου, το διεφθαρμένο σύστημα του Κομμουνιστικού Κόμματος εκείνη την εποχή. Ω μία από τι ακτιβίστριε στο κίνημα, θυμάμαι πολύ καλά πόσο σημαντικό ήταν για μα οποιοδήποτε μήνυμα υποστήριξης και κατανόησης από τη Δημοκρατική Δύση. Σήμερα η πολιτική αντιπολίτευση στη Ρωσία χρειάζεται η νέα γενιά να απαιτήσει τα δικαιώματα της ε, να παγιωθούν στο Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας οι ελευθερία σκέψης, οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Υπερασπιζόμενοι τα βασικά τους δικαιώματα σήμερα παρά της συλλήψεις, ε, τη βία της αστυνομίας ε, πρέπει να συνεχίσουν να αγωνίζονται για το μέλλον της Ρωσίας, μια πιο δημοκρατική Ρωσία που προσέχει περισσότερο τους πολίτες της. Τώρα είναι η ώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξει ότι κατανοούμε και υποστηρίζουμε τα αιτήματα αυτά. Απονέμοντας τον Αλεξέη Ναβάλνη το βραβείο μπορούμε να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα στο ρωσικό λαό και στην αντιπολίτευση ότι πιστεύουμε επίσης πως η Ρωσία μπορεί να είναι πιο δημοκρατική, πιο διαφανής, ε, πιο ευρωπαϊκή χώρα, ότι δεν έχει χαθεί κάθε ελπίδα. Έχω ένα όνειρο να δω τη Ρωσία πιο δημοκρατική. Ίσως όχι στη διάρκεια της δικής μου ζωής, αλλά δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε τα όνειρα για μια δημοκρατική Ρωσία. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Ευχαριστώ. Merci, madame. Chers collègues. Ως γυναίκα, ως ε, μητέρα, συγκινήθηκα ιδιαίτερα από την ε, ε, παρουσίαση της ε, συναδέλφου μας ε, που μας εξήγησε πόσο παρούσα είναι ακόμα η δεκτομή στην Αφρική. Η εφαρμογή ICAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στην Κένια αλλά και σε άλλες χώρες και στην Ευρώπη έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων εκτιμά ότι 16 τουλάχιστον κράτη-μέλη παρουσιάσουν τέτοιου κινδύνους. Παρόμοιε εφαρμογές ε, μπορούν να βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Έχουν ήδη αναπτυχθεί, για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι ε, το 2015. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ομάδα μου θα, το φιλελευθέρων θα ψηφίσει υπέρ αυτού. Ο κ. Αλεξάνδρου Ιορτάνοφ. Ευχαριστώ πολύ. Υποστηρίζω την να βάλει. Γιατί? Γιατί είμαι πεπισμένος ότι είναι ο πιο καλός υποψηφίος. Αν του απονεμηθεί το βραβείο αυτό θα αποτελέσει το πιο ισχυρό και γλαφυρό μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε προς τον ρωσικό λαό. Νομίζω ότι η απονομή του στον κύριο Ναβάλνη θα έχει πραγματικό αντίκτυπο στην Ρωσία αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες. Δυστυχώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να υπάρχουν πολίτες άτομα που ακόμα δεν κατανοούν σε βάθος τις απειλέ τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Τις απειλέ τις οποίες αντιπροσωπεύει το καθεστώ του, του Κρεμλίνου. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε ένα καθημερινό υβριδικό πόλεμο εναντίον μας, εναντίον ε, των αρχών μας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας. Ε, υπάρχουν ασφαλώς πάρα πολλοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Και υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι μεταξύ των υποψηφίων. Όμω ο Αλεξέη Ναβάλνη έχει κάτι παραπάνω. Δεν είναι απλό υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστή. Είναι σύμβολο ελευθερία του λόγου ελευθερία σκέψης. Και έχει ακολούθους, ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτόν. Το είδαμε στο βίντεο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τον παρακολουθούν, που πιστεύουν σε αυτόν. Καθήκον μας είναι να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στο καθεστώς του Κρεμλίνου ότι θέλουμε η Ρωσία να αλλάξει και ότι στο Ναβάλνη βλέπουμε το άτομο που εργάζεται ακούραστα, άοκνα προς αυτή την κατεύθυνση. Περασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ένας ενεργός πολίτης που αναζητεί το καλύτερο μέλλον για τη Ρωσία και τους Ρώσους. Thank you. And the last one is uh, Vladimir. Ευχαριστούμε, Για να είμαι ειλικρινής, ε, έχω μπερδευτεί. Και ηθικά δεν αισθάνομαι άνετα. Για να... Γιατί πρέπει να κάνουμε αυτή την επιλογή που είναι δύσκολη. Ε, λογικό πολιτικό, πολιτικά είναι να επιλέξουμε τον Ναβάλι, είναι προφανές ε, τους, τον ακτιβιστή από την Κίνα. Αλλά κάνοντας κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι αναλαμβάνουμε μια τεράστια ηθική ευθύνη εάν ε, δεν τιμήσουμε τους ηρωικούς Βραζιλιάνους ή τα κορίτσια από την Αφρική. Δεν μπορώ να διανοηθώ να κάνει μια τόσο σκληρή επιλογή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν δίνουμε Όσκαρ εδώ. Δεν βραβεύουμε ταινία ή κοστούμια ή σκηνοθεσία ή σενάριο πρώτο γυναικείο ρόλο είναι πραγματικοί άνθρωποι, είναι πραγματικοί ήρωες και ηρωίδες και πρέπει να τους δείξουμε ότι τους σεβόμαστε, ότι τους γνωρίζουμε, ότι τους θυμόμαστε συνέχεια, ότι τους υποστηρίζουμε, τους υποστηρίζουμε ότι διαμαρτυρόμαστε για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους και για τις δολοφονίες. Δεν ξέρω τους λεπτομερείς κανόνες αυτού του βραβείου, αλλά αν μας επιτρέπουν να δώσουμε πάνω από ένα βραβείο, θα πρέπει να κάνουμε ακριβώς αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν νομίζω ότι ζήτησε καποιο άλλο το λόγο. Κλείνουμε εδώ αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Το είπαμε, ο Μπερνάρ το είπε προηγουμένω, οι άνθρωποι και οι ομάδε ανθρώπων που είδαμε σήμερα στι παρουσιάσει των διαφορών μελών. Όλοι υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν πληρώσει ορισμένοι με τη ζωή τους. Άλλοι με φυλάκιση. Άλλοι εξακολουθούν να αγωνίζονται για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το βραβείο αναγνωρίζει τη δέσμευσή του και τι προσπάθειε του για την υπερασπίση τη ελεύθερη σκέψη με σημαντική επίδραση στη ζωή του, αλλά όχι μόνο στη δική του, προσωπικά, αλλά και στη ζωή τη οικογένεια του των συγγενών. Και αυτό βραβεύουμε εδώ με το βραβείο Ζαχάροφ την προστασία και την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ όλους όσοι παρουσίασαν τις προσωπικότητες αυτές και θα σας παρουσιάσω τη διαδικασία τώρα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα που έχουμε. Το επόμενο βήμα της διαδικασίας του βραβείου Ζαχάροφ θα είναι η ψηφοφορία των τριών επιλαχόντων που έχει προβλεφθεί για την 3η 8 Οκτωβρίου εδώ στις Βρυξέλλες σε μια κοινή συνεδρίαση ΑΦΕΤ ΔΕΒΕ που θα λάβει χώρα και κλεισμένο των θυρών. Η διάσκεψη των Προέδρων τέλος θα καθορίσει το... ποιο θα λάβει το βραβείο από του τρει επιλαχώντε. Όποιο κερδίσει το βραβείο θα κληθεί για μια ανταλλαγή απόψεων σε μια κοινή συνεδρίαση ΑΦΕΤ ΝΤΕΒΕ και ΝΤΡΟΑ τη βράδυ της 16ης Οκτωβρίου στο Στρασβουργό με την, 18 Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου την απονομή του βραβείου. Στη, συγγνώμη, Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο θα υπάρχει η, η εκδήλωση και μετά Τετάρτη 18 θα απονεμηθεί το βραβείο. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.